αναλάβει αύριο. Ευχαριστώ πολύ για το έργο σας και καλωσορίζω την, καλή, την κυρία Γιούροβα. Κύριε Κατάιναν, ευχαριστώ πολύ. Και τώρα φτάνουμε στο επόμενο σημείο, στο επόμενο θέμα μας, δήλωση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενδεχόμενη έκδοση του Τζούλιαν Καλώς Καλωσορίζω Λοιπόν, την κυρία Σιώτα, έχετε το λόγο. Αξιότιμα μέλη, Επίτροπε κυρία Γιούροβα, ευχαριστώ για την ευκαιρία να συζητήσουμε το θέμα της ενδεχόμενης έκδοσης του Julian Assange. Όλοι γνωρίζουμε ότι όταν ενεργεί κανείς για προστασία των ε, δημοσίων συμφερόντων, οι καταγγέλλοντες παίζουν σημαντικό ρόλο για να καταγγέλουν διάφορες ε, παράνομες ενέργειες και γι' αυτό ε, χρήζουν προστασίας νομικής. Το συζητήσαμε αυτό χθε στην συζήτηση που είχαμε για την οδηγία για τους καταγγέλλοντες. Όλοι παρακολουθούσαμε τα πρόσφατα γεγονότα που σχετιζόταν με τον κύριο Ασάνς. Ο Τζούλιαν Ασάνς κατέφυγε στην πρεσβεία του Εκουαδόρ στο Λονδίνο το 2012 για να αποφύγει να απελαθεί στην Σουηδία για να δικαστεί για βιασμό ε, και διάφορα, διάφορες κατηγορίες έλεγε ότι το ήθελε να αποφύγει να εκδοθεί στη ΣΥΠΑ και να δικαστεί γιατί δημοσίευσε χιλιάδες επί χιλιάδων ε, πλαστογραφημένα έγγραφα των ΗΠΑ. Στις 11 Απριλίου το Εκουαδόρ απέσυρε το άσυλο του κυρίου Ασάνς και αυτό οδήγησε στη σύλληψή του από τη Βρετανική αστυνομία. Το δικαστήριο του Westminster ακολούθως τον βρήκε ένοχο για κατηγορίες των Βρετανών για παραβίαση της εγγύηση με την οποία έχει απελευθερωθεί. Πέρα από τι κατηγορίε του Ηνωμένου Βασίλειου, ο κ. αντιμετωπίζει και κατηγορίε και στι ΗΠΑ και οι Σουηδικέ δικαστικέ αρχέ ανέφεραν ότι οι έρευνε που αφορούν το άτομό του ίσω οδηγήσουν να απαγγελθούν εκ νέου κατηγορίε για βιασμό. Να πω ότι το Συμβούλιο αυτό καθε αυτό δεν έχει συζητήσει το ζήτημα του κυρίου Ασάνς και το ενδεχόμενο έκδοσή του και δεν έχει κάποια θέση από αυτού. Είναι γεγονός ότι οι εκδόσεις είναι θέμα αποκλειστικής αρμοδιότητας ε, των κρατών μελών. Γι' αυτό το θέμα τώρα βρίσκεται στα χέρια του Βρετανικού δικαστικού κλάδου και ε, του Υπουργού Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου. Δράτω με τη ευκαιρία όμω να τονίσω εκ νέου ότι το Συμβούλιο προσδίδει πολύ μεγάλη σημασία στην προστασία των κατακέλλοντων είναι γεγονός κατά τη διάρκεια τελευταίου μήνα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εστιάστηκαν επί του, της εξασφαλίσεως συμφωνίας όσον αφορά την οδηγία για τους καταγγέλλοντες και να καταλήξουμε συμφωνία πριν ε, ολοκληρωθεί αυτή η θητεία. Αυτός ο στόχος επετεύχθη και αυτή η Ολομέλεια ψήφισε σήμερα το κείμενο που συμφώνησαν οι διαπραγματευτές των δύο συνομοθετικών κλάδων. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ για αυτά που μας είπατε, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον λόγο τώρα έχει η κυρία Γιούροβα εξ ονόματος της Κομισιόν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας ζήτησε να κάνουμε μία δήλωση για την πιθανή έκδοση του Τζούλιαν Ασάντζ από το Ηνωμένο Βασίλειο. Μπορούμε να σας ενημερώσουμε πως η έκδοση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών ε, βασίζεται σε διμερή συνθήκη και Συμφωνία Έκδοσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν επιτρέπεται η έκδοση στην περίπτωση που υπάρχουν λόγοι να υποψιαζόμαστε, να θεωρούμε ότι μπορεί να υπάρξει εφαρμογή της ανατικής ποινής. Επιπλέον λέγεται πως το κράτος μέλος δεν θα πρέπει να προχωρήσει σε έκδοση εάν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων του υπόπτου στην περίπτωση που η Σουηδία αποφασίσει να εκδώσει νέο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης μετά από αυτό το οποίο είχε ανακαλέσει το 2017 και το Βρετανικό Δικαστήριο θα έπρεπε να εξετάσει το εάν θα προηγηθεί το ε, ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης ή το αμερικανικό ένταλμα έκδοσης. Δεν υπάρχουν σαφείς κανόνες, αλλά κάποιοι παράγοντες που θα λάβει υπόψη το δικαστήριο. Ως γενική παρατήρηση πρέπει να σημειώσω πως η Κομισιόν δεν έχει αρμοδιότητα για να παρέμβει σε δικαστικές διαδικασίες που εκκρεμούν στα δικαστήρια των κρατών μελών. Βασιζόμαστε πλήρω στην ανεξαρτησία και τον επαγγελματισμό των Βρετανικών δικαστηρίων για να λάβουν την σωστή απόφαση, ε, καθώς έχουν και μπροστά τους τα στοιχεία. Σας ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο πρώτος ομιλητής είναι ο κύριος Πόσπισιλ για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να συμφωνήσω ε, με την Επίτροπο και να πω και εγώ ότι δεν καταλαβαίνω γιατί συζητούμε την υπόθεση αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε μια συγκεκριμένη υπόθεση αιτήματο έκδοσης που θα εκδικαστεί με βάση τις διεθνείς συμφωνίες. Έχουμε την δικαιοδοσία του Ηνωμένου Βασιλείου, έχουμε τις Ηνωμένε Πολιτείε που ζητούν την έκδοση. Πρόκειται για δύο κράτη δικαίου και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η δικαστική διαδικασία θα είναι απόλυτα σωστή με τις κατάλληλες οικονομικές ε, εγγυήσεις και με σεβασμό του κράτους δικαίου. Μπορούμε να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε με τις ενέργειες του κ. Ασάνζ. Εγώ διαφωνώ. Θεωρώ ότι η ελευθερία έκφρασης έχει τα όρια του και δεν μπορεί να, και να παραβιάζει το ε, απόρριτο, το εθνικό ή τους όρους εθνικής ασφάλειας. Αλλά Σίγουρα οι αρμόδιες δικαιοδοσίες θα πρέπει να αποφασίσουν για την υπόθεση Ασάνς και είναι σωστό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι οι πολιτικές αρχές δεν δικαιούνται να επεμβαίνουν στο δικαστικό σύστημα, στη δικαστική εξουσία μιας άλλης χώρας. Ας αφήσουμε το ζήτημα στα Βρετανικά δικαστήρια, στους Βρετανούς δικαστές που θα εκδικάσουν το αίτημα της έκδοσης και θα κρίνουν αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την έκδοση του κυρίου Ασάνς στις Ηνωμένε Πολιτείε. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο Βρετανικό δικαστικό σύστημα. Ευχαριστώ κυρία Γκόμες εκ μέρους Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Η έκδοση του ζηλίας σας προς τις Ηνωμένες ε, θα πρέπει να παρεμποδιστεί. Μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε ε, προστασία της Ευρώπης όποιον θέλει διαφάνεια και, προσ... και ε, προασπίζει την αλήθεια όταν μια κυβέρνηση σαν το Τραμπ που, που χρησιμοποιεί τα ΜΜΕ για τους δικούς στόχους δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε την έκδοση του Ασάνς ε, γιατί ο κύριος Τραμπ ε, έχει εργαλειοποιήσει αυτό το θέμα ε, και ο Ασάνς θα διέτρεχε κίνδυνο να καταδικαστεί ακόμη και στην ασχάτη των ποινών όπως επισημαίνουν σημαντικές οργανώσεις ε, πίεσης, ε, ε, προστασίας δικαιωμάτων. Είδαμε τι έγινε με την περίπτωση του Μάνικ που υπέστη και βασανιστήρια για την καταγγελία κάποιων στοιχείων. Είδαμε τι έγινε στο Γουαντάναμο και στις μυστικές φυλακές. Είναι τρομερή η υποκρισία των Αμερικανών και των συνένοχων μερικές φορές ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Και μάλιστα ένας υπουργός που με καταδίκασε όταν ζήτησα διερευνητική ε, επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να εξετάσουμε τις μυστικές πτήσεις ε, ε, στην Πορτογαλία και σε μυστικές φυλακές από το Γουαντάναμο, με κατηγόρησαν ότι προσπίζω τον ιδρυτή του Wikileaks. Το Wikileaks. Θα πρέπει λοιπόν αν όντως διέπραξε κάποια αδικήματα ο κύριος Ασάνζ να δώσει λόγο στα σουδικά δικαστήρια που δίνουν τις δικονομικές εγγύσεις για τη δίκαιη δίκη αλλά να μην γίνει η έκδοσή του προς τις Ηνωμένε Πολιτείε. Με ανησυχεί ιδιαίτερος που ε, ο Ζούλιαν Ασάνζ παραδόθηκε από την ε, πρεσβεία του ησημερινού από μια χώρα που συνεργάστηκε με τον Πούτιν για να επέμβει στις αμερικανικές εκλογές. Και είδαμε τι έγινε με την ειδική περίπτωση του Μίλλερ στις Ηνωμένε Πολιτείε. Θα πρέπει λοιπόν να εγγυηθούμε δικαιοσύνη και δίκαιη δίκη στον Ζουλιαν Ασάνζ. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τον Ασάνζ, να προστατεύσουμε τους ε, καταγγέλλοντες και να εγγυηθούμε τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες. Ε, να προστατεύσουμε αυτούς που διακινδυνεύουν τη ζωή τους για την ελευθερία και τη διαφάνεια. Ο Ζουλία Σάνζ αξίζει την προστασία μας και αξίζει να απολαύσει όλα αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δέχεστε μια γαλάζια κάρτα από τον κύριο Πόσπισιλ. Κύριε Πόσπιση, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφε, παρακολούθησα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ε, την παρέμβασή σα. Είμαι πρώην Υπουργό τη Δικαιοσύνη και σα ερωτώ το εξή. Πώ είναι δυνατό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομοθετική εξουσία να επεμβαίνει σε μια δικαστική υπόθεση. Μιλούμε για μια διαδικασία έκδοσης ε, ε, είναι μια υπόθεση που απασχολεί τα δικαστήρια. Εμεί είμαστε πολιτικοί. Δεν μπορούμε να προστατεύουμε εμεί ως πολιτικοί ε, κάποιον όπω ε, προτείνατε, κάποιον που ενέχεται σε μια διαδικασία έκδοση. Πώς το δικαιολογείτε. Κοιτάξτε, δεν πρέπει καμία ευρωπαϊκή χώρα να κάνει εκδόσει προ μια χώρα που έχει τη θανατική ποινή και αυτό ισχύει για τι Ηνωμένες και λυπάμαι γι' αυτό. Και πράγματι ο Ασάντ, αν εκδοθεί στι Ηνωμένε Πολιτείε, μπορεί να μετωπίσει κατηγορία για κατασκοπία που συνεπάγεται θανατική ποινή. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ε, νομικό και πολιτικό λόγο για τον οποίο δεν πρέπει να εκδοθεί από ένα δικαστήριο είτε στον Ηνωμένο Βασίλειο, είτε στη Σουηδία, είτε στη δική σα χώρα. Σα ευχαριστώ πολύ. Επόμενο, ο κ. Ουρμπαν Κρέσπο, εκ μέρου τη ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ. Η κράτηση του Ασάνς σηματοδοτεί μια πολύ σκοτεινή στιγμή για την ελευθερία της έκφρασης. Η σύλληψη και κράτησή του μας ε, αγγίζει όλους και τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν χάρη στον Ασάνς και το Wikileaks ε, αποκάλυψαν δολοφονίες δημοσιογράφων, ε, πολλοί άριθμες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο και η ομάδα εργασίας για τις αυθαίρετες κρατήσεις κρέκρινε παράνομη την κράτηση του Ζούλια Ρασάνς. Επίσης, έχουμε κρούσει το κόδωρο του κινδύνου για την έκδοση του ΑΣΑ στις ε, Ηνωμένε Πολιτείε. Σήμερα εγκρίναμε οδηγία για την προστασία των πληροφοριοδοτών. Θα πρέπει να την τηρήσουμε. Η έκδοση του ΑΣΑ θα έδινε ένα πολύ επικίνδυνο μήνυμα. Θα έδινε το μήνυμα ότι αυτοί που υψώνουν το παράστημά τους ε, απέναντι στη διαφθορά, στην κατάχρηση εξουσία το πληρώνουν με το κεφάλι του αν τον εκδώσουμε στι Ηνωμένε Πολιτείε, ουσιαστικά θα απαρνηθούμε θεμελιώδη τιμά τη δημοκρατία μα. Θα απαρνηθούμε το αναπαλωτρίο, το δικαίωμα στην ελευθερία έκφραση. Α μην το επιτρέψουμε, κυρίε και κύριοι. Σα ευχαριστώ. Τον λόγο έχει η κυρία Εύα Ζολή. Η ενδεχόμενη έκδοση του Ζούλιαν Ασάνς, του ιδρυτού του Wikileaks, προ τι Ηνωμένε Πολιτείε, είναι κάτι που δεν αφορά τη μοίρα ενό ανθρώπου, αλλά σκιαγραφούμε έτσι και το μέλλον των δημοκρατιών μας. Θα πρέπει να επερασπιστούμε με κάθε προσπάθεια την ελευθερία τη ενημέρωση, τη πληροφόρηση και τη διαφάνεια, διότι περί αυτού πρόκειται. Ο Ασάντ δημοσιοποίησε πληροφορίε που ανησυχούν, ταράσουν, κυρίω για εγκλήματα πολέμου που διεπράχθησαν από τι ΗΠΑ. Παρά να λάβουμε υπόψη το έγκλημα, να λάβουμε υπόψη το έγκλημα, η κυβέρνηση θέλει να αποσιωπήσει, να σιωπήσουν οι φωνέ που ακούγονται. Θα πρέπει να ενταχθούμε σε αυτό. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τη δημοκρατία την ανοιχτή, τη διαφανή, ε, και να είναι υπεύθυνε οι πράξεις μας. Το θάρρος του είναι αυτό που κρίνεται σήμερα. Εάν δεχθούμε να εκδοθεί ο Ασάνς, θα εκδώσουμε αύριο όλους εκείνους που δημοσιεύουν πληροφορίες ευαίσθητες, δημοσιογράφους του Guardian, της Moon, του Spiegel, που δημοσίευσαν έγγραφα ε, που έχουν βρει από το Wikileaks η Γαλλία, θα πρέπει να δώσει άσυλο στο Julian Assange και να υπερασπιστεί το χρώμα της διαφάνειας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, εκ μέρους του EFTD, το λόγο έχει ο William Dartmouth. Ευχαριστώ. Ας ξεκινήσουμε με μία πρόταση, μία αρχή. Δεν είναι καλή ιδέα οι πολιτικοί να προσπαθήσουν να παρέμβουν σε μία νομική διαδικασία. Αυτό πραγματικά είναι μία πολύ κακή ιδέα ο διαχωρισμός πολιτικής και νόμου είναι στο επίκεντρο των αξιών της Δυτικής Δημοκρατίας. Στην περίπτωση του κυρίου Τζούλιαν Ασάνς ε, συνελήφθη ε, προσήχθη στο δικαστήριο και καταδικάστηκε διότι θεωρήθηκε ότι ήταν ένοχος ε, παραβίασε τις συνθήκες εγγύησης. Είναι διαφορετικέ οι κατηγορίε του Χάκιν και άλλε παρεμφερεί κατηγορίε που τα παγκέθηκαν στι ΗΠΑ. Αυτέ είναι τα αντικείμενα τη ακρόση περί εκδόσεω. Η ακρόση θα λάβει χώρα ενώπιον δικαστού Βρετανού. Και αυτό που είπε το Συμβούλιο ήταν από τα γεγονότα ασφαλμένο. Ο Υπουργό Εσωτερικών δεν είναι αυτό που αποφασίζει. Πολλοί, εμού συμπεριλαμβανομένου, ε, διαφωνούσαν με κάποιε αποφάσει δικαστών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά κανένα σοβαρό άνθρωπο αμφισβητεί την αντικειμενικότητα και τον επαγγελματισμό του αγγλικού δικαστικού κλάδου. Παρόλα αυτά, η κυρία Γκόμεζ και άλλοι συνάδελφοι θέλουν η νομική αυτή διαδικασία να υπόκειται σε πολιτική παρέμβαση. Αυτή είναι η τελευταία μου ομιλία στο Κοινοβούλιο και πρέπει να διαφωνήσω. Το να συζητάμε, ε, να εξαρτούμε, να επηρεάζουμε πολιτικά τη δικαστική διαδικασία είναι κάτι που είναι αντίθετο όχι μόνο στι δυτικέ αξίε, αλλά κυρία Ζολή, εναντίον όλων των θεσμών τη δημοκρατία. Θα πρέπει εμεί ω πολιτικοί να αφήσουμε το θέμα, το νομικό θέμα του Τζούλιαν Ασάνζ στην ησυχία του, να μην το αγγίξουμε. Τώρα, ποιε ήταν οι αρχικέ νομικέ διαδικασίε που οδήγησαν στο να ξεφύγει, να παραβεί τι συνθήκε για την εγγύησή του, του κ. Σάντ, ήταν το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη. Και αυτό το ένταλμα σύλληψη δεν εκδόθηκε από Σουηδό δικαστή, αλλά από Σουηδό εισαγγελέα. Παρά τα αυτά, με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης δεν υπάρχει πραγματική υπεράσπιση κατά της έκδοσης. Και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Ακούμε πολλά εδώ περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άρα το, οι σοσιαλιστές, οι φιλελεύθεροι, οι Βρετανοί φιλελεύθεροι, όλοι οι υποστηριχτές του ευρωπαϊκού υπερκράτους που δεν σκέφτονται καν, είναι οι ίδιοι άνθρωποι εκείνοι που είναι μεγάλοι υποστηρικτές του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Οι προσπάθειες που κατέβαλαν για την προστασία πολιτικών δικαιωμάτων και για το ευρωπαϊκό εντάλμα σύλληψης είναι πολύ ασφαλμένες προσπάθειες, όπως και στην περίπτωση του κυρίου η προσπάθεια που καταβάλατε για προστασία πολιτικής ελευθερίας και για σωστές νομικές διαδικασίες κολλάνε στο καλέ. Και όλα εν ονόματι ε, μεγαλύτερης ολοκλήρωσης. Εάν αυτοί οι άνθρωποι σκεφτόταν, ξανασκεφτόταν, σας εκλυπαρώ, σας παρακαλώ να το ξανασκεφτείτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Τέλειος Κούλογλου από την ΚΟΕ έχει το λόγο. Άκουσα δύο πόντιους πιλάτους ε, σήμερα. Είμαστε υπέρ ε, των καταγγελόντων, αλλά δεν έχουμε αρμοδιότητες. Το Συμβούλιο και η Κομισιόν. Εδώ πέρα όμως είμαστε εμείς πολιτικό σώμα. Μπορούμε να έχουμε μια πολιτική άποψη για τα γεγονότα. Ακούστε τι γίνεται. Ας υποθέσουμε ότι ένας Ευρωπαίος δημοσιογράφος γράφει κάτι ή κάνει μια αποκάλυψη ε, για το Ιράν. Εάν ο Ασάνς εκδοθεί, υπάρχει ένα προηγούμενο εδώ. Δηλαδή, το Ιράν θα μπορέσει να ζητήσει έκδοση του δημοσιογράφου αυτού ή η τουρκια Ή ε, να τον συλλάβει ή να τον απάγει. Ε, τι θα πείτε τότε. επειδή λέει παραβίασε ε, τα, τα μυστικά του Ιράν, της Τουρκίας ή οτιδήποτε. Μην παίζετε τον Ποντιο Πιλάτο λοιπόν εδώ πέρα. Όταν κινδυνεύει η ελεύθερη πληροφόρηση και σταυρώνονται οι ε, καταγγέλλοντες. Σας ευχαριστώ. Υπάρχει μια μπλε κάρτα από την Άννα Γκόμες. Την δέχεστε, ναι. Σας ευχαριστώ. Κύριε Γκόμες. Συμφωνώ με τον συνάδελφο Είμαστε πολιτικό σώμα και μπορούμε να εκφέρουμε πολιτική κρίση. Και αυτό κάνουμε. Λέμε δεν πρέπει να εκδοθεί στη ΣΥΠΑ. Από την άλλη, αναμένουμε τα δικαστήρια στο Ηνωμένο Βασίλειο που ευτυχώς ε, θα παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να δεσμεύονται από την Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τις ε, συνθήκες και άρα υπάρχει κάποια νομική και όχι πολιτική βάση για να μην υπάρξει έκδοση σε μια χώρα που έχει ακόμα θανατική ποινή. Συμφωνείτε κύριε to Συμφωνώ πλήρως. Πρέπει να κάνουμε μια δήλωση. Έχουμε κάνει δηλώσεις επιδηλώσεων για τη Βενεζουέλα, την Τουρκία, για ε, ε, ε, τα πάντα. Και ο συναδελφός μου εκεί πέρα μιλάει για νομική διαδικασία. Έγινε σεβαστή η νομική διαδικασία στην περίπτωση άλλων χωρών. Κάνουμε παρεμβάσεις, δηλώσεις. Γιατί όχι τώρα. Επειδή είναι σε αυτό το χάλι η Βρετανική κυβέρνηση λόγω Brexit και προσπαθεί να ξεμπλέξει με τον αντιπερισσοσμό του εσά. Δεν είναι σωστό Όχι. Είστε πολιτικό, πρέπει να λάβετε μία θέση. Είστε υπέρ ή κατά τη έκδοση. Σα ευχαριστώ. Ε, Βεβαίω, ε, ερωτηθήκατε, έχετε δικαίωμα να απαντήσετε. Κυρία Πρόεδρε, ε, χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία να απαντήσω. Είναι νομικό ζήτημα. Αυτό είναι. Τελεία και παύλα. Λοιπόν, τώρα, εάν είστε υπέρ του οι πολιτικοί να παρεμβαίνουν στις δικαστικές διαδικασίες, είναι κάτι το κατανοητό και θεμητό. Αλλά εγώ ε, δεν συμφωνώ. Αλλά είναι δικαίωμά σας να το υποστηρίζετε αυτό. Αλλά είναι τελείως αντίθετο με τον τρόπο που ε, λειτουργούν οι δυτικές δημοκρατίες η διάκριση της εκτελεστικής από τη δικαστική εξουσία είναι θεμελιώδης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άννα Μιράντα για ένα λεπτό, εκ μέρους των Πρασίνων. Ένα λεπτό σας δίνω το λόγο. Θα σας ρωτήσω το εξής, συνάδελφε. Τι γίνεται με τις δίκες στην ε, Τουρκία. Η Τουρκία σωστά λέει ότι αυτό είναι νομικό ζήτημα, νομική, νόμιμη δράση και ότι πρέπει να σεβαστούμε τη, νόμιμη, τη νομική διαδικασία στην Τουρκία και να μην παρέμβουμε. Τότε γιατί εμείς κάναμε τόσες δηλώσεις κατά δικών στην Τουρκία. Γιατί. I Ρητορικό το θεωρώ το ερώτημα. Επιθυμείτε να απαντήσετε. Όχι, ναι. Να απαντήσω σε μερικά δευτερόλεπτα. Αυτό που προτείνει, διατείνεται ο συνάδελφος, είναι ότι η Βρετανική κυβέρνηση θα έπρεπε να παρέμβει σε μια δικαστική διαδικασία στην Αγγλία. Αυτό που λέτε για την Τουρκία είναι να παρέμβετε ή να επιδιώξουμε να παρέμβουμε στην Τουρκία. Συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ με τις επικρίσεις κατά της Τουρκίας. Και μακάρι η κυβέρνησή μου και άλλες κυβερνήσεις να καταστήσουν σαφέ ότι η Τουρκία ποτέ δεν θα γίνει μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανεξάρτητα κατά πόσο το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι μέλο ή όχι. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Και οι δύο πλευρέ ακούστηκαν. Θα μπορούσατε να πιάσετε μεγάλη κουβέντα. Α δώσουμε το λόγο στην επόμενη συνάδελφα, Άννα Μιράντα από του Πρασίνου. Ευχαριστώ πολύ. Την ε, Δευτέρα είχα ραντεβού με τον ε, Ζουλένα Σάνς ε, στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο. Δεν πήγε γιατί στο μεταξύ συνελήφθη. Παραβιάστηκε το δικαίωμά του σε άσυλο και φυλακίστηκε. Ε, το δικαίωμα του ασύλου σημαίνει προστασία από την θανατική ποινή και απόλυτη προστασία δικαιωμάτων. Το άσυλο που ζήτησε ο Ασάζ είναι για να προστατευτεί από την ε, ηλεκτρική καρέκλα και να προστατευτεί το δικαίωμα της ελευθεροτυπίας σε μια χώρα που δεν θα είχε δικαίωμα σε δική δίκη. Ε, Παρ' όλα αυτά παραβιάστηκε το δικαίωμα ασύλου του Ζουλιάν Ασάνζ και παραβιάστηκαν τα δικαιώματά του. Έγιναν δεκτές ε, δεκάδες δίκη ε, ε, καταδίκη ε, στις Αμερικανικές φυλακές. Η Βρετανική κυβέρνηση δεν απαιτεί εγγύηση από τις ΗΠΑ για να μην εφαρμογεί της θανατικής ποινής, γιατί στις επιστολές που βρέθηκαν στο, στο στην, ε, στην Υπουργή Δικαιοσύνη του Ισημερινού διαπιστώνουμε ότι δεν έχουν αναλυθεί ούτε εγγυήσει ούτε υποσχέσει να μην εκδοθεί ο Ζουλιάν στις στι Πολιτείε. Το Ηνωμένο Βασίλειο ουδέποτε δεν έδωσε εγγύηση για μη έκδοση. Και θεωρούμε ότι ο σημερινός με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο συντονίστηκαν για να συλλάβουν τον Ασάνζ. Δεν θα πρέπει να εκδοθεί ε, ο Ασάνζ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα γίνει κάτι τέτοιο οποιοδήποτε δημοσιογράφος που ε, καταγγέλει διαφθορά ή κατάχρηση εξουσίας θα μπορεί να έχει την ίδια μοίρα. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Η κυρία Κονέτσνα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σήμερα ψηφίσαμε μία οδηγία όπου προβλέπεται η προστασία εκείνων που καταγγέλουν ε, διάφορα γεγονότα και να τους προστατεύουμε. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε αυτό. Αυτό ψηφίσαμε σήμερα. Σε αυτή την έκθεση και σχετικά με αυτό θα ήθελα να πω ότι όλα τα μεγάλα σκάνδαλα που αποκαλύφθηκαν ε, τελευταία όπως τα LuxLeaks ή τα Panama Papers Όλα αυτά αποκαλύφθηκαν χάρη σε καταγγέλλοντε. Ήταν προ το δημόσιο συμφέρον. Έτσι δεν είναι. Δεν με νοιάζει πραγματικά. Δεν με νοιάζει αν η Ασάσα Ζούλια Ασάντ είναι προδότη είναι ήρωα. Ε, τον θεωρώ σε αυτή τη φάση αυτό το γεγονό δευτερευού τη σημασία. Αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό είναι ότι αν θέλουμε να προστατεύουμε του καταγγέλλοντε, πρέπει να προστατεύσουμε τον Ασάντ. Θα πρέπει να εκδοθεί προ μια χώρα στην οποία ο πρόεδρος θεωρεί το δημοσιογράφο σαν έναν εχθρό του λαού. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι μια τέτοια δικαιοδοσία θα είναι δίκαιη σε μια τέτοια χώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το λόγο έχει η Επίτροπος η κυρία Γιούροβα. Έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση που είχαμε. Θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που είπα προηγουμένως. Εμείς ε, ε, υπολογίζουμε πλήρως στην ανεξαρτησία και τον επαγγελματισμό των Βρετανικών δικαστηρίων. Και πιστεύω ακράδαντα ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα και το δικαίωμα για δίκαιη δύση θα γίνουν πλήρως σεβαστά στις αποφάσεις των Βρετανικών δικαστηρίων. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει εκπρόσωπος τη Ρουμανικής Προεδρίας, η Υπουργός Τσιότ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επιτρόπε, κυρίες και κύριοι, για να ολοκληρώσουμε. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για την ε, ευκαιρία που μου δώσετε να συζητήσουμε αυτό το επίκαιρο ζήτημα και θα, να σας ευχαριστήσω που συζητήσατε αυτό το θέμα της υπόθεσης Ζουλιάνα Σάνς και ευχαριστώ για την προσοχή. Το ολοκληρώθηκε η συζήτηση, τελείωσε και η ημερήσια διάταξή μας. Θα συνεχίσουμε το έργο μας αύριο στις 8.30 αύριο το πρωί. Έχει δημοσιοποιηθεί η ατζέντα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η σε διάταξη. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ για τη δουλειά που κάνατε. Γεια σας.